Ja, Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die Plätze ein. Wir haben gestern Χθες, αγαπητοί συνάδελφοι, αποφασίσαμε να τροποποιήσουμε την ημερησία διάταξη και έχουμε το 15 υπαριθμών 15 έκθεση δηλαδή για την ανάπτυξη, επικύρωση και νομική αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων που μπορούν να υποκαταστήσουν τις δοκιμές σε ζώα στον τομέα των καλλιντικών. Και θα ακολουθήσει το 16 προφορική ερώτηση της Μαργκρέτε Άουκεν σχετικά με την αναβολή αναθεώρησης του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας στο είδωρο. Από τις 10 και 40, 11 παρά 20, θα αρχίσουμε να ψηφίζουμε τα 10, 13, 14, 11 και μετά για τα ε, καύσιμα στην αυτιλία, τα ναυτικά καύσιμα. Θα αρχίσω λοιπόν τώρα το, τη συζήτηση του υπαριθμών 15 αλλά θα δώσω πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Α, η οποία είναι παρούσα, βεβαίω. Η κυρία Σμινό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα στις κυρίες και τους κυρίους Ευρωβουλευτές. Η τελευταία έκθεση που δημοσιεύσαμε για τα καλλιντικά και για τις δοκιμές σε ζώα. Όπως γνωρίζετε, η σχετική οδηγία προβλέπει σταδιακή κατάργηση των πειραμάτων σε ζώα για καλλιτικά. Μια τέτοια απαγόρευση ισχύει ήδη από το 2004 για την απαγόρευση πειραμάτων επί των συστατικών και συνδυασμών συστατικών από το 2009. Και από το Μάιο του 2009 απαγορεύεται επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση η διάθεση στην εμπορία καλλιτικών και συστατικών τα οποία έχουν δοκιμαστεί επιζών. Αυτή η απαγόρευση διαθέσεως στο εμπόριο απαγορεύεται, απαγορεύει τη χρήση των συστατικών προϊόντων, ε, κρατικών προϊόντων και υπάρχει προθεσμία του Μαρτίου του 2013. και ε, ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά. Η οδηγία προβλέπει ότι στην περίπτωση όπου υπάρχουν εναλλακτικέ επιλογές στις δοκιμασίες επιζών θα πρέπει εφόσον δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα μέχρι το 2013, θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα καταθέσει νομοθετική πρόταση. Κατέθεσε η Κομισιόν την ε, πρότασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τις εναλλακτικέ δυνατότητες ε, τον Σεπτέμβριο του 2011 με διπλό σκοπό αφενός για να ικανοποιήσει τα προβλεπόμενα από την οδηγία περικαλυτικών, από την άλλη για να ενημερώσει τα δύο άλλα θεσμικά όργανα ότι η κατάσταση των animal tests δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί πριν από τις 11 Μαρτίου 2013 χωρίς να προκαταλαμβάνει στην έκθεσή της το πώς θα αντιμετωπίσει την έλλειψη εναλλακτικών επιλογών στα πειράματα σε ζώα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά η προοπτική είναι θετική. Αν εξετάσει κανεί τι εξελίξει από το 2003, όταν δηλαδή άρχισε η εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων. Τα τεστ σε ζώα ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Ο αριθμός πειραματοζώων έχει μειωθεί στον αριθμό 344 που αυτός ήταν ο τελευταίος αριθμός του 2009 πριν να καταργηθεί απολύτως. Έχει γίνει πρόοδος και στη διεθνή συνεργασία όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για την αξιολόγηση μεθόδων στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για τις ρυθμίσεις για τα καλλιτικά. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι σημαντικοί πόροι διατέθηκαν και εξακολουθούν να διατίθενται για την έρευνα με συνολικό ποσό χρηματοδότησης μεταξύ 2007 και 2011 στα 200 περίπου, 100, ε, στα 200 περίπου εκατομμύρια από τα οποία 42 εκατομμύρια για την αξιολόγηση και πρόθεση εναλλακτικών προγραμμάτων. Η βιομηχανία καλλιτικών παίζει ενεργό ρόλο στη συμβολή στην προσπάθεια αυτή με ανάληψη δραστηριοτήτων έρευνας καθώς και με συγχρηματοδότηση όπως για παράδειγμα τα 25 εκατομμύρια που διέθεσε ο κλάδος σε ένα κοινό project στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Σε ό,τι αφορά την διαθεσιμότητα εναλλακτικών μεθόδων για την προθεσμία του 2009, ε, βελτιώνονται οι μέθοδοι για την έλεγχο, για τον έλεγχο της τοξικότητας και γίνεται πρόοδος. Ανεξαρτήτως της προθεσμίας του 2013 και των σημαντικών προσπαθειών που γίνονται στην έρευνα, η αξιολόγηση και κατοχύρωση εναλλακτικών μεθόδων δεν θα είναι εξασφαλισμένη πριν από την έναρξη της απαγόρευσης. Γνωρίζει την κρίσιμη σημασία της διαθεσιμότητας εναλλακτικών μεθόδων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2013. Και στη σύνταξη της εκθέσεως που τίθεται υποσυζήτηση σήμερα, δεν βασίστηκε μόνο στις δικές της γνώσεις, αλλά αναζήτησε και τη διαβούλευση με τρίτα μέρη, με τους ενδιαφερόμενους, με τη βιομηχανία, με μη κρατικούς οργανισμούς, καθώς και με τις χώρες μέλη και με την επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με την προστασία των καταναλωτών. Από όλους αυτούς ζητήθηκαν, ζητήθηκε εμπειρογνωμοσύνη. Αναλύθηκαν οι σχετικές μελέτες από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αξιολόγηση Αναλλακτικών Μεθόδων έκανε και δημόσια διαβούλευση το 2010 επί του σχεδίου εκθέσεως που είχαν συντάξει οι εμπειρογνώμονες. Με τίτλο «Εναλλακτικές μέθοδοι έρευνας μη βασιζόμενες σε πειραματόζα» και μπορούν να βρεθούν αυτά και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης έχουν δημοσιευθεί και στο επίσημο έντυπο. Και σε, σε έχουν, και σε ε, ε, έντυπα. Το, οι διατάξει του 2003 έδειχναν καθαρά ότι θα είναι πολύ δύσκολο να εξευρεθούν εναλλακτικέ μέθοδοι. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να επανεξετάσει την κατάσταση πριν από το 2013. Επίσης, στην ετήσια έκθεση τα τελευταία έτη, στις ετήσιες εκθέσεις μάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε κατ' επανάληψη τις δυσκολίες στην εξέβρεση εναλλακτικών μεθόδων που να αντικαταστήσουν τα πειραματόζωα. Για τα επόμενα βήματα τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της κατάστασης στην έκθεσή της για την προστασία των ζώων, για την ασφάλεια των καλλιτικών που είναι διαθέσιμα στου καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο, για το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Η απαγόρευση εμπορίας, εφόσον δεν υπάρχουν αλλακτικέ μέθοδοι, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην δυνατότητα να εισαχθούν στην αγορά νέα συστατικά καλλιτικών καθώς επίσης και, να χρησιμο... και, τη τη χρησιμοποίηση υφιστάμενων στατικών. Ακόμα δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για το πώς η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Όπως ίσως γνωρίζετε, η Κομισιόν βρίσκεται σε διαρκή επαφή με πολλούς από τους ενδιαφερόμενους για το θέμα αυτό. Και εκτός από τις επιλογές που έχω εξηγήσει από την αρχή, δηλαδή διατήρησης της προθεσμίας ή αναβολής. Συζητείται τώρα μάλιστα και ένας αριθμός άλλων στοιχείων, εκ των οποίων ένα είναι να μην υπάρξει αναβολή της προθεσμίας, αλλά να χορηγούνται εξαιρέσεις αναπερίπτωση για την είσοδο στην αγορά ορισμένων συστατικών, βεβαίως υπό την τήρηση αυστηρών όρων. Η δέσμη μέτρων θα επιτρέπει θα επιτρέπεται χρήση υπορισμένου όρου υφιστάμενου στρατικών. Και βεβαίω ε, θα γίνεται η αξιολόγηση και ούτω καθεξή. Για την διατήρηση υψηλού επίπεδου προστασία των ζώων. Επιτρέποντα ωστόσο την πρόσβαση των καταναλωτών σε νέα σημαντικά προϊόντα που θα προσφέρουν τη προστιθέμενη αξία μέσω του μηχανισμού των εξαιρέσεων. Αυτό ίσως αποτελεί τη βάση για μια εξισορροπημένη προσέγγιση και να προσφέρει κίνητρα για την διεξαγωγή έρευνας, αν και δεν θα αποκόψει την Ευρωπαϊκή Ένωση απολύτως από την καινοτομία στον χώρο των καλλιτικών. Yeah an äh, Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ορισμένοι έχουν ήδη εγγραφεί στον κατάλογο των αγορητών. Όπως θα προσέξατε έχουμε επισκέπτες από το Βερολίνο. Η ομάδα που έχει προσκαλέσει η Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ και καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Μέλη της Europarty σωματίου, δηλαδή, εγκεκριμένου σωματίου, και πρώτη θα λάβει το λόγο βέβαια η Dagmar Ροτ Μπέρεντ, η οποία είχε αναλάβει παλαιότερα την εισήγηση του σχετικού θέματος και μετά θα ακολουθήσουν άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε θα εξηγήσω στους ε, καλεσμένους μου γιατί δεν μιλώ γερμανικά. Θα μπορούσα να μιλήσω γερμανικά, θα με μετέφραζαν τέλεια οι συνάδελφοι, μου, οι συνάδελφοι μάλλον της ε, γερμανικής καμπίνας και ίσως και θα προτιμούσα να το έκανα, να μίλαγα γερμανικά, αλλά για να είναι πιο άμεση η επαφή με την ε, εκπρόσωπο της Επιτροπής, την κυρία Λεγκρινιέ, θα μιλήσω αγγλικά. Αλλά Βερολινέζοι, να είστε σίγουροι, εδώ μιλάμε και γερμανικά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πράγματι ε, για οποιαδήποτε σχετική με τα καλλιντικά νομοθεσία τα τελευταία, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, 17 χρόνια ήμουν εισηγήτρια. Τώρα δεν ξέρω τι περιμένει από εμά η Κομισιόν. Πράγματι υπήρχαν τρία ανοιχτά τελικά σημεία. Πράγματι υπήρχε η προθεσμία για τον Μάρτιο του 2013. Ναι, είναι προφανέ ότι αυτή την προθεσμία δεν τη χρειαζόμαστε. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα λοιπόν. Εγώ ως εισηγήτρια που Προασπίζομαι ε, να σταματήσουν τα πειράματα στα ζώα για μια νέα οδοντόκραμη, δεν ξέρω εγώ τι, να, πει, να πω ότι ναι, είναι πολύ ευαίσθητο, πολύ λεπτό θέμα και ε, επιτρέπεται να βρεθούν διάφορες λύσεις. Εγώ να πω ότι σέβομαι και κατανοώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το οποίο περιμένετε εσείς από εμά. Ίσως και εμείς κατά το παρελθόν θα έπρεπε να είχαμε δραστηριοποιηθεί περισσότερο παρότι από τον κλάδο έχω ακούσει ότι για κάποια endpoints, για κάποια τελικά σημεία δεν υπάρχουν και πολλές δυνατότητες. Πάντοτε στρέφομαι σε ανθρώπους που έχουν περισσότερες επιστημονικές γνώσεις από εμένα. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου και γι' αυτό θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική και να μην δώσω την εντύπωση ότι είμαι έτοιμη να ενδώσω σε αποδυνάμωση της νομοθεσίας. Αλλά αυτό το οποίο ε, θέλω να δώσω ως ε, τροφή για μελέτη στην κυρία Λεγκρινιέ και θα περιμένω και την απάντησή της είναι το εξής. Το πρώτο πράγμα, αν βρούμε ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες για αυτά τα τρία endpoints μέχρι τον Μάρτιο του 2013, αν γίνει αυτό, το πρώτο που μπορώ να πω εγώ είναι ένα ερώτημα. Τα χρειαζόμαστε και αυτά τα τρία τελικά σημεία για όλα τα καλλιντικά. Ο επιστημονικός ε, κόσμος ε, ε, έχει κάποιες απόψεις. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουμε καταλήξει και στα τρία αυτά τα τελικά σημεία. Γι' αυτό σας παρακαλώ λοιπόν να κάνετε τη διάκριση με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και να μας πείτε ποια είναι τα πρώτα για τα οποία δεν χρειαζόμαστε αυτά τα endpoints. Και ολοκληρώνω όπου να είναι κύριε Πρόεδρε. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι όταν έχουμε κάνει αυτή τη διάκριση Αυτά που είπατε εσείς, δεν θέλω να το παρουσιάσω ως δική μου ιδέα, αλλά σας ρωτάει εσάς κύριε Αλεγκρινιέ. Αυτό που είπατε, ε, μιλήσατε για κάποιες εξαιρέσεις και κάποιες κατά περίπτωση. Ε, ξέρεις, τι, γιατί μιλάμε, για νέες ουσίες, εντελώς νέες ουσίες, για τις οποίες θα υπήρχε εξαίρεση και για τις οποίες θα υπήρχε τεράστια αξία ε, για τον πληθυσμό. Και αυτή την αξία ποιος θα την πει, ποιος θα την καθορίσει, μια επιτροπή δεντολογίας ηθικής, και σε ό,τι αφορά την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων από όλα πλαίσια, τι πιστεύετε, αν μια ουσία έχει ε, χρησιμοποιηθεί, ε, έχει δοκιμαστεί ως χημικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να δοκιμαστεί πάνω σε ζώα, μήπως έχουμε κάποια και πώς θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε αυτό. Και σε λίγο θα ξαναπάρω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ε, Μετρώ πέντε συναδέλφους που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο. Κανονικά θα έπρεπε να είχα πει στην κυρία Ροτμπέρεντ ήδη μόνο 1,5 λεπτό ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε όλου του συναδέλφου και να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ πάντω όλε και όλου από εδώ και πέρα 1,5 λεπτό. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο, αλλά για να είμαστε δίκαιοι και απέναντι στου άλλου και να μπορέσουμε να ακούσουμε όλου όσοι επιθυμούν να μιλήσουν και να αρχίσουμε την ψηφοφορία στι 10.40. Η κυρία Ρωμάνα Ζόρνταν Σίσελη και μετά θα ακολουθήσουν άλλες και άλλοι συνάδελφοι. Um, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση προβλέπει τώρα δηλαδή απαγόρευση για το 2013. Από την άλλη μεριά έχουμε τους εμπειρογνώμονες και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται πως δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε όλα ε, τα πειράματα σε ζώα. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά την πολιτική και τα λόγια που λέει και από την άλλη μεριά έχουμε την πραγματικότητα. Και το 2013 είναι μεθαύριο. Αν λοιπόν εμείνουμε στην απαγόρευση και μας οδηγήσει αυτό στην εισαγωγή α, καλλιτικών προϊόντων, τότε θέτουμε σε κίνδυνο την ε, υγεία των προϊόντων και ούτω ή άλλω θα είναι και λιγότερα τα προϊόντα που θα είναι διαθέσιμα στην αγορά. Η εξέλιξη νέων προϊόντων βελτιώνει την ασφάλεια των καταναλωτών. Μακροπρόθεσμα λοιπόν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας και βεβαίως λιγότερο ασφαλή σε σύγκριση με άλλα που προέρχονται από άλλα μέρη του κόσμου. Και βεβαίως αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο και με ανησυχεί είναι η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Και δεν μιλώ μόνο για τις μεγάλες ε, βιομηχανίες, μιλώ και για μικρές και μεσές επιχειρήσεις, για την ασφάλεια των θέσεων απασχολήσεως και ε, σε περίοδο κρίσεως πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα πριν να θεσπίσουμε τέτοια νομοθετήματα. Λοιπόν, νομίζω ότι το να επιτραπούν εξαιρέσεις είναι αναπόφευκτο. Ε, αλλιώς ε, θα είναι ε, η κατάσταση ε, βλαβερή για όλους. Τα χρήματα επίσης για τις έρευνες είναι πολύ σημαντικά. Πολλά χρήματα έχουν δοθεί για την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων. Πρέπει να βρούμε ένα μοντέλο το οποίο να μην ενθαρρύνει τη βιομηχανία να μην αναζητεί εναλλακτικές μεθόδους. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή για τη δήλωσή της. Να συγχαρώ την Επιτροπή και τη βιομηχανία των καλλιντικών και τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις για τα βήματα προόδου την τελευταία δεκαετία, σημαντικά βήματα προόδου. Χαίρομαι που δεν έκανε και κάποιες επιπλέον συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα απαιτούσαν από πλευράς μας απόκριση τεχνικής επάρκειας Κατανοούμε την πραγματικότητα βέβαια. Βλέπουμε ότι πριν 10 χρόνια είχαμε κάνει δηλώσεις λέγοντας ότι δεν θα πρέπει εμείς να επιβάλλουμε πόνο στα ζώα για να, για να αποκτήσουμε νέα προϊόντα που θα εξυπηρετήσουν αποκλειστικά την ανθρώπινη ματαιοδοξία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να αποσυρθεί κανένα από τα προϊόντα τα οποία είναι ήδη στην αγορά. Έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα και θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχει εξετάσει τις εναλλακτικέ λύσεις που προτείνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις σχετικά με τα τεστ, τα οποία τα πειράματα και τα τεστ, τις δοκιμασίες εκεί όπου δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης των ζώων από των πειραματοζώων από άλλες μεθόδους. εφόσον διεκδικήσουμε την άμεση και πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ε, ακούγονται απειλές για απώλεια εκατοντάδων ή χιλιάδων θέσεων εργασίας. Ας μας πει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συμβαίνει. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα επιτρέψουμε περιπτωσιακά εξαιρέσεις αν δούμε κατάλληλη ε, προστιθέμενη αξία. Να μας εξηγήσει τι σημαίνει πράγματι σημαντική προστιθέμενη αξία. Τι εννοεί με αυτό. Η κυρία Γκροστέτ και μετά ο Ρώση. Ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα θέμα που έχουμε επανειλημμένα συζητήσει. Να θυμίσουμε ότι η βιομηχανία των καλλιντικών είναι από τις πλέον καινοτόμους βιομηχανία στην Ευρώπη. Η ηγέτης του τομέα της στον κόσμο η ευρωπαϊκή βιομηχανία παράγει πολύ, έχει θέσεις απασχόλησης υψηλού επίπεδου, συνεργάζεται με πολλά ερευνητικά ιδρύματα και θυμίζω ότι δεν υπάρχουν μόνο μεγάλες βιομηχανίες, υπάρχουν χιλιάδες μικρομεσαίες ιδιαίτερα δυναμικές. Είναι πρωτοπόρος, πρόδρομος της μεθόδους ε, τεστ και ελέγχου των νέων ουσιών και προϊόντων και όχι μόνο με ζώα, έχει μεσολαβήσει και η δράση δική μας που οδήγησε την βιομηχανία να χρησιμοποιεί και άλλες μεθόδους, να βρει άλλες μεθόδους οι οποίες είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν για να αποδειχθεί το μη βλαπτικό του προϊόντος τους πριν από την κυκλοφορία στην αγορά. Τώρα, οι πειραματισμοί με πειραματόζωα για την μη τοξικότητα των ουσιών δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο εάν υπάρχει εκ των προτέρων έγκριση. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για πράγματα που πρέπει να ολοκληρωθούν διαδικασίες μέχρι τον Μάρτιο του 2013, πολύ σύντομα δηλαδή. Οπότε τι γίνεται. Θα υπάρξουν προϊόντα τα οποία θα απαγορευθούν ενώ είναι ιδιαίτερα κατάλληλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δει ποσοτικά σε επίπεδο θα έλεγα βιομηχανίας και έρευνας και μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν διατηρήσει αυτή την ημερομηνία του 2013 πόσα πειραματόζωα θα σώσει. Ο κύριος Ορέστε Ρώση. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ευαίσθητα όλα αυτά τα θέματα και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να δώσουμε τον απαιτούμενο χρόνο στην Επιτροπή για να λάβει τα σωστά μέτρα. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες θα έλεγα στη δική μας Επιτροπή. Θα ήθελα κάτι το πιο συγκεκριμένο. Εμείς είμαστε, θα έλεγα, καταδικασμένοι να παρατείνουμε ουσιαστικά τις αδειοδοτήσεις για χρήση πειραματοζώων. Θέλουμε όμως εγγυήσεις για να το κάνουμε αυτό. Πρώτον, να μην υπάρχει υποχρεωτική χρήση των ζώων και να μην υφίσταται η δυνατότητα αυτή για το σύνολο των καλλιντικών προϊόντων. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να απαγορεύσει την εμπορία και την εισαγωγή από τρίτες χώρες προϊόντων καλλιντικών τα οποία προβλέπουν ακόμα και για ένα τμήμα τους μόνο ε, την χρήση πειραματοζώων. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαληθεύσει έτσι ώστε τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες δεν περιλαμβάνουν συστατικά τα οποία έχουν γίνει αντικείμενο πειραματισμού σε ζώα. Λοιπόν, από τη μία ναι στην απαγόρευση θα έλεγα των πειραμάτων με ζώα αλλά ναι στον αυστηρό έλεγχο των εισαγωμένων προϊόντων και του τρόπου με τον οποίο έχουν εγκριθεί. Ζανόνι. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που συμβαδίζει με την κοινή γνώμη την Ευρωπαϊκή σχετικά με τους ελέγχους των καλλιντικών προϊόντων. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θέλει να πει όταν λέγει εδώ ότι δεν θέλει να ξεπεραστεί η προθεσμία η χρονική, αλλά θα δοθούν κατ' εξαίρεση κατά περίπτωση άδειες και για τους ελέγχους. Οι έλεγχοι από ποιου θα γίνονται, από τα κράτη-μέλη ή υπάρχει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός για την τέλεση αυτών των ελέγχων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο νομίζω έτσι ώστε οι κανονισμοί και οι οδηγίες να εφαρμόζονται και να εφαρμόζονται σωστά. Αν αρχίσουμε τώρα να δίνουμε και εξαιρέσεις ε, δεν είναι καθόλου σωστό και γι' αυτό θα πρέπει να παραμείνει η χρονική προθεσμία του Μαρτίου 13 η κυρία Οκονή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ όπως και όλοι σας είμαι φυσικά υπέρ ε, της απαγόρευσης των πειραμάτων σε ζώα στον τομέα της βιομηχανίας των καλλιντικών, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Πρώτα απ' όλα είμαι υπέρ της προστασίας των καταναλωτών. Η απαγόρευση των πειραμάτων δεν νομίζω ότι θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ποιοτικά τα πειράματα που γίνονται, άρα αυτό να υπονομεύσει την προστασία των καταναλωτών που όλοι έχουμε ως προτεραιότητα στην Επιτροπή μας. Και αν υπάρχει τέτοιο κίνδυνος αυτό πρέπει να το δούμε. Χθε στην ε, Σύνοδο Κορυφής οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων έκαναν ε, το δυνατό για να προτείνουν σχέδια ανάπτυξη, ε, σχέδια συνδεδεμένα με την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μα. Εκ παραλίου, λοιπόν και εμεί πρέπει να επαγρυπνήσουμε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι μεν να βαδίσουν προ την κατεύθυνση τη απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα, αλλά όχι με οδήποτε τίμημα. Η Φρανσουά Γκροστέτ μας θύμισε κάποια αριθμιστικά στοιχεία για τη βιομηχανία καλλιντικών πόσο σημασία έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τη δυνατότητα να βρούμε κάποιες άλλες αναλλακτικέ επιλογές. Και πρέπει να έχουμε χρόνο για να το κάνουμε. Ξέρουμε ότι μπορούν να μετεγκατασταθούν αυτές οι βιομηχανίες και δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την ε, μετεγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό. Mm. Έχω μια παρατήρηση προς την Κομισιόν ε, και μετά θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ε, η ερώτησή μου προς την εκπρόσωπο την Κομισιόν είναι αν έχετε αριθμητικά στοιχεία. Μπορείτε να μας πείτε πόσα πειράματα σε ζώα μπορέσαμε να αποφύγουμε. Φαντάζομαι ότι εδώ μιλάμε για λίγο πολύ επώδυνα πειράματα και δοκιμές. Θέλω να μας μιλήσετε και για το αντίστοιχο ποσοστό άπαξ και εφαρμοστεί η νέα ε, νομοθεσία. Οι συνάδελφοι, συνάδελφοι από το ΕΛΚ μας είπαν ότι πρέπει να δούμε λίγο πιο σχετικά το ζήτημα της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής. Αλλά ξέρετε, δεν ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε. Υπάρχει ήδη και συμφωνώ με τον Κρίς Ντέιβις. Εδώ δεν μιλάμε για την ασφάλεια του καταναλωτή, διότι αυτή έχει ήδη εξασφαλιστεί. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι σε ποιο βαθμό μπορούμε να επιτρέψουμε να υποφέρουν ζώα για να έχουμε πιο πολλά κραγιόν σε πιο πολλά χρώματα. Υπάρχουν προϊόντα αναγνωρισμένα εγκεκριμένα, αρκετά τον αριθμό. Μέχρι πού θέλουμε να φτάσουμε, αφού γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες. Κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να αναγνωριστούν, δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί. Και σίγουρα Υπάρχουν πολύπλοκες διαδικασίες για να αναγνωριστούν αυτές οι συναλλακτικέ. Υπάρχει και ένα intergroup για την καλή μεταχείριση των ζώνων. Είμαι πρόεδρο αυτή τη ομάδα αυτή τη στιγμή. Και είναι θέματα αυτά που μας απασχολούν εδώ και χρόνια. Πάντως δεν πρέπει να κάνουμε στροφή 180 μοιρών και να δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα. Καρ Σλούτερ. Υπάρχουν δεκάδε χιλιάδε ουσίε που μπορούν να συνδυαστούν και να δημιουργήσουν εκατοντάς χιλιάδε νέα καλλιντικά δεν είναι θέμα ασφαλής, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε χημικά και δεν πρέπει να κάνουμε καμία εξαίρεση. Άλλωστε, είναι μια από τις νομοθεσίες που γνωρίζει, τις ελάχιστες που γνωρίζει ο πρέπει Πολίτης και είναι πολύ ικανοποιημένο με τις διατάξεις αυτής της νομοθεσίας. Όχι ευχαριστούμε λοιπόν καμία παράταση, κανένα νέο, καμία νέα χημική ουσία, καμία εξαίρεση. Κανένα πείραμα στα ζώα. Είναι σαφή η νομοθεσία δεν πρέπει να αλλάξει. 29 δευτερόλεπτα. Συμπληρωματική ερώτηση από την κυρία Ροτ Μπέρεντ. Επανέρχομαι στην κυρία Λεγκρινιέ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή. Μπορεί η κυρία Λεγκρινιέ να μας πει, διότι ένα πράγμα πρέπει να πω. Αν θέλουμε να εμείνουμε στην προθεσμία, πρέπει να εμείνουμε στην προθεσμία. Έχουμε την ίδια ιστορία με τις στοιχείες κλοβών ορνήθων, όπου τα αυγά από τις συστοιχίες αυτές εξακολουθούν να φτάνουν στην αγορά παρόλο που απαγορεύονται εδώ και μια δωδεκαετία. Όπως είπε και ο Κριστέβης, όπως είπα και εγώ, πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στα προϊόντα εκείνα τα οποία δεν χρησιμοποιούν τα συστατικά που έρχονται από πειραματόζωα κτλ. Και να πούμε αυτά, ανάμεσα αυτά και στα άλλα. Και να εφαρμόσουμε την προθεσμία και αν χρειαστεί να πάμε και στα δικαστήρια. Να πάτε εσείς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν, αν είναι δυνατόν, συντομότατα διότι έχουμε ήδη καθυστερήσει πολύ. Έχουμε άλλωστε ένα θέμα ακόμη να συζητήσουμε. Η κυρία Λεγκρενιέ πρέπει να πάει σε άλλη συνάντηση και γι' αυτό θα την αντικαταστήσω. Έπρεπε έτσι και αλλιώ να ήμουν από την αρχή εδώ, αλλά χρειάστηκε η κυρία Λεγκρενιέ να είναι σέσιμο. Δύο πολύ σημαντικά θέματα να υπογραμμίσω. Πρώτον, Νομίζω ότι αυτό που μας απασχολεί κυρίως είναι η προσπάθεια διασφάλισης, θα έλεγα, των καταναλωτών, των καλλιντικών προϊόντων. Δεν υπάρχει καμία παραχωρητικότητα σχέση με αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν είναι αρκετά δεδομένα διαθέσιμα για την εγγύηση των προϊόντων αυτών, δεν θα αδειοδοτηθούν και αν τεθούν ερωτήσεις για την ασφάλεια μιας κάποιας ουσίας η οποία ήδη χρησιμοποιείται και αν δεν υπάρχουν δεδομένα για να τεκμηριώσουν τη χρήση της, τότε τα προϊόντα θα πρέπει να αποσυρθούν. Πρώτον ήταν αυτό. Δεύτερον, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα δεν έχει πάρει καμία απόφαση για το τι θα κάνει σε σχέση με την υπάρχουσα τεκμηρίωση. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες. Η πρώτη, να επιτρέψουμε την προθεσμία να τεθεί σε ισχύ χωρίς τροπολογήσεις και χωρίς καθυστερήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, όπως είπα, η νομοθετική ρύθμιση είναι ήδη έτοιμη. Οι άλλες δυνατότητες που προσφέρονται σήμερα είτε είναι να αναβληθεί η χρονική στιγμή ή η διατήρηση της χρονικής στιγμής με κάποια δυνατότητα εξαιρέσεων και στις δύο αυτές περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις οι οποίες θα έρθουν προς έγκριση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Είπατε αν χρειάζονται όλα τα endpoints για όλα τα προϊόντα. Όχι, αλλά αυτά τα οποία ζητούνται είναι τεστ γενικότερα τοξικότητας και τοξικότητας δερματικής ή δερματολογικής καλύτερα. Και στην περίπτωση αυτή ζητείται να γίνουν έλεγχοι όπου τα τεστ δεν είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματά τους. Για τις άδειε τώρα, τις εξαιρεσει. για να υπάρξουν εξαιρεσει θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες μόνο για αυτούς οι οποίοι τις χρειάζονται. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμες οι εξαιρέσεις αυτές όπου υπάρχει πραγματικά σημαντική προστιθέμενη αξία από τη χρήση των νέων ουσιών. Σαν παράδειγμα, κάποια συντηρητικές ουσίες δείχνουν ότι είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές βακτηριολογικά, ως εκ τούτου θα υπάρξουν μέτρα. Δεν θα δοθούν εξαιρέσεις μόνο και μόνο γιατί τα νέα συστατικά που προτείνονται οφείλονται στο ότι μπορούν να παραχθούν με χαμηλότερο κόστος ή ε, είναι απαραίτητα για να υπάρξει σαν παράδειγμα ένα νέο χρώμα για κραγιόν. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρόκειται να ε, δοθεί εξαίρεση. Η εξαίρεση μπορεί να ζητηθεί από έναν μεμονωμένο κατασκευαστή ή από ένωση κατασκευαστών. Θα πρέπει να αποδείξουν ο ένας ή ο άλλος ε, τα δεδομένα τοξικότητας ε, τα οποία δεν ήταν μέχρι τότε διαθέσιμα και δεν μπορούν να τα πετύχουν με εναλλακτικέ μεθόδους. Θα πρέπει να δώσουν διασφαλίσεις για τα τεστ επιζώων που θα πρέπει να γίνουν και κάτω από ποιες συνθήκες. Και θα πρέπει επίσης να δείξουν ότι θα επενδύσουν προς αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων ελέγχου. Λοιπόν αυτή είναι η λογική γύρω από τις εξαιρεσει. θα πρέπει η λογική αυτή να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, δεν έχουμε καταλήξει σε μια τελική διατύπωση. Απαντώντας τώρα στην ερώτηση του ότι δεν θα επηρεαστούν τα προϊόντα της αγοράς. Κοιτάξτε, αν τεθούν προβλήματα ασφαλείας, τότε κάποια προϊόντα πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά ή μπορεί να αποσυρθούν. Έχουμε κάποια δεδομένα για τις επιπτώσεις στη βιομηχανία, στην περίπτωση επίσης εφαρμογής των ρυθμίσεων, επιπτώσεις στην απασχόληση, στην έρευνα, στην καινοτομία. Έχουμε περάσει στη φάση μιας μελέτης επιπτώσεων, και θα είναι διαθέσιμη όταν ολοκληρωθεί στα μέλη του Κοινοβουλίου. Για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Οι εισαγωγές των καλλιντικών προϊόντων ένας εισαγωγέας πρέπει να καταθέσει ένα τεχνικό φάκελο που να δίνει εγγυήσει για την ασφάλεια των προϊόντων ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που είναι ισχύει στην περίπτωση των προϊόντων που κατασκευάζονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει να είναι οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στο φάκελο αυτό παραπλανητική για τα τεστ σε ζώα. Τον προηγούμενο χρόνο έγιναν 1500 τέτοια τεστ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν κάνω λάθος τα περισσότερα από τα τεστ αυτά έγιναν σε ε, ποντικούς και αρουραίους κυρίως, σε μικρά τροκτικά. Το 2009, τον προηγούμενο χρόνο που είχαμε, εν πάση περιπτώσει, ήταν αρκετά νόμιμο να χρησιμοποιηθεί, είχαν γίνει 344 τέτοια τεστ, οπότε ε, βλέπετε ε, την, ε, τις συνέπειες της διαφοράς ανάμεσα στους αριθμούς. Ελπίζω να απάντησα. Ο Πρόεδρος, Ευχαριστώ. Προχωρώ αμέσως στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως, την προφορική δηλαδή ερώτηση για το θέμα του νερού. Και θα παρακαλέσω πολύ σύντομα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί για τρία λεπτά. Και μετά ένα λεπτό η κυρία Άουκεν και μετά πάλι συντομότατα θα μπορέσει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν, έχουμε δυνατότητα να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Η Κομισιόν λοιπόν σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Όκεν για την προφορική της ερώτηση. Με πολύ μεγάλη χαρά σας ανακοινώνω ότι από σήμερα 10 η ώρα το πρωί έχει εγκριθεί επίσημα η πρόταση από την Κομισιόν. Είναι μια πρόταση που οποία καθυστέρησε κάπως, αλλά όπως γνωρίζετε οι αποφάσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνονται σε συλλογική βάση. Κάποιες φορές ένας ε, επίτροπος μπορεί να θέσει κάποιες ερωτήσεις σε κάποιον άλλο. Εσωτερικά λοιπόν χρειαζόμαστε χρόνο για να δοθούν οι απαντήσεις. Πάντως τώρα έχουμε την πρόταση αυτή στη διάθεσή μας. Δεύτερο τμήμα, αν υπήρξε σημαντική αλλαγή του σχεδίου πρότασης της Κομισιόν. Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή στις ε, προτάσεις της Κομισιόν. Η πρόταση αυτή είναι στο πλαίσιο τη οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Στόχο έχει τη ρύθμιση των χημικών ουσιών. Υπάρχει ήδη οδηγία του 2008 η σχετική και πρόκειται για επικαιροποίηση της ε, εν λόγω οδηγία ε, με προσθήκη 15 νέων ουσιών στον ε, κατάλογο των ουσιών για τι οποίε υπάρχουν οριακές τιμέ που θα πρέπει να σέβονται τα κράτη-μέλη. Περιλαμβάνονται σε αυτές τις ουσίες ουσίες που, είναι, που έχουν να κάνουν με ε, ζυζανιοκτώνα, βιοκτώνα, ε, βιομηχανικά, χημικά. Έχουν να κάνουν με ενδοκρινική διαταραχή, κάποιους παράγοντες ε, και κάποιες άλλες ουσίες και άλλη καινοτομία του κανονισμού αυτού. Είναι δημιουργία μιας watch list ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κομισιόν πολλές φορές όταν εκπονεί τέτοιου είδους προτάσεις είναι η έλλειψη δεδομένων, ένα είδος φαύλου κύκλου. Υπάρχουν ε, υποχρεώσει να παρακολουθούνται κάποιε ουσίε, αλλά αυτέ οι ουσίε είναι ήδη καταγεγραμμένε. Το θέμα είναι να πάρουμε πληροφορίε για να προωθήσουμε αποφάσει συμπερίληψη νέων ουσιών στου υφιστάμενου καταλόγου. Θα δημιουργηθεί λοιπόν ένα ad hoc κατάλογο για την παρακολούθηση, τον έλεγχο για μια διετία περίπου και εν συνεχεία οι πληροφορίες αυτές που θα έχουμε συγκεντρώσει θα χρησιμοποιούνται για την ε, ενδεχόμενη προσθήκη νέων ουσιών σε αυτόν τον κατάλογο. Δεν ξέρω αν ε, ξεπέρασα τα 2,5 λεπτά, αλλά νομίζω ότι σας έδωσα σε αυτό το διάστημα τα ουσιώδη στοιχεία της πρότασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό παρακαλώ κύριε Άουκεν. Και μετά για άλλο ένα λεπτό ο κύριος Ζέμπερ. πολύ. Θα σας μιλήσω στα δανέζικα σήμερα, γιατί μπορώ, επειδή και οι δύο είμαστε δανείοι εκπρόσωπος Κομισιόν και εγώ, να μιλήσουμε πιο άμεσα. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο περιμένω με την απάντηση αυτή. Χαίρομαι πάρα πολύ με όλα όσα μας είπε ο εκπρόσωπος Κομισιόν. Ένα ερώτημα προς σαν εκπρόσωπο αυτό. Αυτό το ερώτημα είναι το εξή. Μπορεί η Κομισιόν να λάβει υπόψη τι δυνατότητε του άρθρου 16 παράγραφος 8 Μπορείτε να μας διατυπώσετε συγκεκριμένες προτάσεις για να ξέρουμε ακριβώς τι μπορεί να γίνει στην πράξη. ότι γνωρίζω ότι σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν αρκετές αοριστείες. Αν θέλουμε όμως να υπάρχει διαφάνεια, θα πρέπει να ε, περάσουμε το μεσόρο, να βάλουμε πιο ψηλά τον πύχη. Θα πρέπει η Κομισιόν λοιπόν να παρέμει προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί λοιπόν η Κομισιόν να μας ε, διαβεβαιώσει ότι θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες στο άρθρο 16 εδάφιο 8. Είχε διατυπωθεί η νομοθετική πρόταση ε, το 1990, αλλά τελικά αποδυναμώθηκε εντελώ. Μήπως πρέπει να αποκαταστήσουμε ε, κάποια κομμάτια αυτής της πρότασης του 1990. Ο κ. Ζέμπερ, ευχαριστώ. Πρόκειται για σημαντικό θέμα της ημερησίας διατάξεως και θα σας παρακαλούσα στην ε, διάρκεια της συζητήσεως να μην επιτρέπετε στους συναδέλφους να μιλούν δύο φορές, γιατί και χθε το ίδιο κάνατε. Νομίζω ότι όλοι εδώ πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και να καθορίζετε από πριν τον χρόνο αγορεύσεως, όχι να επιτρέπετε σε ορισμένου να, να μιλήσουν για πέντε λεπτά έστω και αν έχουν πολλά πράγματα και ανεξαρτήτως βεβαίω κομματική ε, τοποθετήσεως. Πρόκειται για πρόταση νομοθετική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως και για έκθεση η οποία ενδεχομένω να καταλήξει σε νομοθετική πρόταση. Παρακαλώ λοιπόν ως Πρόεδρος να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και να προσφέρετε την ίδια δυνατότητα να ομιλήσουν όλοι. Τώρα, προς την Επιτροπή. Όπως είπε και ο κ. Τάβιτοφ, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν έχουμε επαρκή δεδομένα σε ό,τι αφορά αυτά τα κατά συστατικά. Πώς θα διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα περιληφθούν στις λίστες και τα νέα ενδεχόμενα επικίνδυνα συστατικά. Για παράδειγμα και υπόλοιπα, η κατάλοιπα μάλλον φαρμάκων. Στην Ελβετία για παράδειγμα έχει μπει και μια τέταρτη διαδικασία φιλτραρίσματος των νερών η οποία δεν υπάρχει στην ε, Ευρώπη, στην ε, Ενωμένη Ευρώπη δηλαδή. Και αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί στο μέλλον. Πρόεδρο, Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Κύριε Ζέμπερ, ακολουθεί η Κομισιόν για να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητήσουμε την υλοποίηση. Νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε την υλοποίηση άπαξ και εγκρίθηκε η πρόταση. Έχει υπάρξει κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τα χημικά μετά την έγκριση της οδηγίας πλαίσια για τα ύδατα. Μετά ήρθε το REACH, ε, είχαμε τους κανονισμούς ε, για τα ζυζανιοκτώνα και τα βιοκτώνα. Άρα και επιπρόσθετα εργαλεία για να έχουμε τα μέτρα τα οποία χρειάζονται αν θέλουμε να φτάσουμε στα πρότυπα που προβλέπονται από αυτήν την οδηγία πλαίσιο. Επίσης υπάρχουν και ε, τα μέτρα που υιοθετούν τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας. Αν δείτε παραδείγματος χάρη κάποια από ε, τα, τις φαρμακευτικές ουσίες δεν υπάρχει πρόβλημα με τα ύδατα όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής αλλά σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Υπάρχουν και προληπτικά μέτρα και διορθωτικά μέτρα, κάποια επεξεργασία των υδάτων, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Κατά περίπτωση, ό,τι αφορά ε, καθοδήγηση δημοσίευση κάποιων κατευθυντήριων γραμμάτων των Κομισιόν έχουν μια κοινή στρατηγική μαζί με τα κράτη-μέλη. Εκεί συζητούμε και τα περί της υλοποίηση της οδηγίας πλαισίου, ποιε είναι οι οδηγίες που μπορούμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη και το καθεξής. Και βεβαίως ε, θα αναφερθούμε στα κράτη-μέλη και για το ενδεχόμενο να υπάρχει ανάγκη δημοσίευση νέων κατευθυντήριων γραμμών. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ζέιμπερ, ε, η ιδέα με αυτό το watch list που θέλουμε να εκπονήσουμε είναι να βάλουμε σε αυτόν τον κατάλογο κάποιες ουσίες και να δούμε κατά πόσον δημιουργούν πρόβλημα, κίνδυνο. Και θα λάβουμε υπόψη μας ε, τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσουμε για μια μελλοντική πρόταση. Κάθε τέσσερα χρόνια είναι η προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων στον τομέα αυτό. Η Κομισιόν θα μπορεί λοιπόν να βάλει τις ουσίες ε, αυτές σε ένα watch list μέσω κατεξουσιοδότησης πράξης, θα τις παρακολουθεί για ένα-δύο χρόνια και μετά τα αποτελέσματα της παρακολούθησης του monitor να τα χρησιμοποιεί ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία λήψεως αποφάσεων ε, για μελλοντικέ προτάσεις ε, και για την καλύτερη υλοποίηση των προτάσεων σε ό,τι αφορά την νέων ουσιών. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, σίγουρα γίνονται πολλά πράγματα στα κράτη-μέλη και με τις φαρμακοβιομηχανίες και σε ό,τι αφορά την ε, θεραπευτική αντιμετώπιση στα νοσοκομεία, την επεξεργασία των λιμάτων ε, στην Ελβετία. Ε, πράγματι υπάρχει ένας κανονισμός ο οποίος θεσπίστηκε και θεσπίζει πρότυπα για κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες και κάποια φαρμακευτικές ουσίες για την κατεργασία που πρέπει να γίνεται στην Ελβετία σε κάποιες ουσίες. Αυτό θα μπορούσαμε ίσως να το υιοθετήσουμε και εμείς στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Ζητώ συγγνώμη που ήταν ε, δυστυχώς σύντομος ο χρόνος που μπόρεσα να σας διαθέσω. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Ελπίζω ότι έχετε όλοι τις κάρτες σας και όπως είπα θα αρχίσουμε με το θέμα υπαριθμών 10. Έχουμε αρχίσει ψηφοφορία όμως. Ορίστε. Ορίστε παρακαλώ. Κύριε, Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικό παρακαλώ. Σύμφωνα με τον κανόνα 156 του εσωτερικού μας κανονισμού, μια τροπολογία μπορεί να ετολογηθεί, να εξηγηθεί από το συντάκτη της και με βάση επίσης τον κανόνα 196 της, ε, του κανονισμού. Ο κανόνας 156 ισχύει για τις ε, επιτροπή. επιτροπής. Σε ό,τι αφορά ε, τον ε, κανονισμό ΣΕΦ, εγώ είχα θέσει χθε το ερώτημα κατά πόσο συζητήσαμε τι τροπολογίε. Οι συντάκτε έχουν δικαίωμα να συζητηθούν οι τροπολογίε. Και δεν είναι ένα δικαίωμα το οποίο μπορεί κανεί να το παραβιάσει. Σας ερωτώ λοιπόν, συζητήσαμε αυτές τις τροπολογίες. Κοιτάξτε, ε, συζητούμε τώρα ε, ένα θέμα το οποίο θα ψηφίσουμε. Για το 88 παράγραφος 2. Γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό σε αυτό Καλά, μιλάτε για άλλο θέμα τη ημερησία διατάξεως. Όταν θα φτάσουμε εκεί, σας παρακαλώ να ζητήσετε ξανά το λόγο. Θα προχωρήσουμε τώρα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ, έχετε όλοι τις κάρτες σας, ψήφι υπέρ. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ψηφίζει με μία ψήφο παραπάνω από ό,τι επιτρέπεται κανονικά. Πέραση της ψηφοφορίας. 45 υπέρ, 15 κατά και 3 άποχες. Το 13 τώρα, η φορολόγηση της ενέργειας. Τροπολογία 58 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, άρα γίνει επαλήθευση γίνει παντήθεση για την 57 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ένα μέλος παραπάνω πάλι οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. ...15 υπέρ 48 κατά... ...απορρίπτεται... ...59 υπέρ... ...κατά... Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Καλά. Για την 7 λοιπόν. Το Λαϊκό Κόμμα έχει τώρα δύο ψήφου παραπάνω. Πέρας, 31 ψήφοι υπέρ, 30 κατά. Εγκρίνεται και καλά που κάναμε την ηλεκτρονική επαλήθευση. ...61 και 62 ψηφίζονται μαζί. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές και εδώ παρακαλώ να γίνει επαλήθευση πέρας 36 υπέρ, 26 κατά, εγκρίνεται. Ενοποιημένη τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές ας γίνει επαλήθευση παρακαλώ 71 πέρας 37 υπέρ 26 κατά 0 αποχές 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά άποχες ας γίνει πάλι και εδώ η παλήθευση. 63 Πέρας. 36 υπέρ, 26 κατά, καμία εποχή. αποχή αλφα υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 65 και 66 υπέρ, κατά, Αποχές. Επαλήθευση της 65 66. Ονομαστική ψηφοφορία δηλαδή. Πέρας. 31 ψήφοι υπέρ και 29 κατά, κατά και 0 αποχές. 67 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69 υπέρ και 69 και 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αυτή τροπολογίες 11, 24 και 8β υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές δεν είναι όμως σαφές το αποτέλεσμα νομίζω ας κάνουμε λοιπόν ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 14 δύο παραπάνω πάλι οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Πέρας. 39 υπέρ 24 κατά εγκρίνεται επομένως. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ενοποιημένη 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Η 15 έχει αποσυρθεί. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Προτιμώ να γίνει μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Abstimmung Ψήφι 38 υπέρ, 24 κατά. ...77 και 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ενοποιημένη 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται αυτή. Θέλετε επαλήθευση. Καλώς. Επαλήθευση λοιπόν για την 79. Ψηφίσατε. 39 ψήφοι υπέρ, 23 κατά εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέλετε επαλήθευση επαλήθευση 81 Πέρας. 35 υπέρ, 24 κατά εγκρίνεται επομένως. Η υπαριθμόν 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται αυτή. Ακολουθεί η 82 και 83 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 84 και 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 και 86 είναι ταυτόσημες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται και αυτή. 90 και 91. Είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Παράρτημα. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 92 και 93 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 94 υπέρ κατά απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα η εισαγωγική έκθεση, οι ιδεολογικές σκέψεις, 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή, 32 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 τέσσερα υπέρ. Κατά. Άποχες. Θα κάνω επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. 34. Πέρας. 32 υπέρ. 28 κατά. Εγκρίνεται επομένω. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 36 υπέρ. Κατά. αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Καλά, θέλετε επαλήθευση λοιπόν. 36. Πέρας. Δύο ψήφοι βλέπω παραπάνω του Λαϊκού Κόμματος. 16 υπέρ 46 κατά. Είναι πάντως σαφές ότι απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές Δεν είμαι βέβαιος. Ας κάνουμε παρήθευση. 38. Πέρας τώρα της ψηφοφορίας, 34 υπέρ, 26 κατά, εγκρίνεται επομένως. Και προχωρούμε στην 40 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 41 και 42 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 2 παρελθόν 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνονται 44 και 48 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτονται. Ναι. Ψηφίζομαι λοιπόν την 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρότιμο να κάνουμε παρήθευση. 49 λοιπόν. Πέρας. 32 υπέρ. 31 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 4 υπάρχουν τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές προτιμώ να γίνει επαλήθευση 52 λοιπόν πέρας 32 υπέρ 30 κατά Εγκρίνεται λοιπόν. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 και 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Υπαριθμόν 6 καθώς και 56 μαζί υπέρ κατά αποχές. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ο συνασπισμός που διαγράφεται. Ας επαληθεύσουμε όμως. 56. Πέρα. 48. Υπέρ 15. Κατά. Εγκρίνεται επομένως. 55. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και μένει ορίστε παρακαλώ η κυρία Βαν ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε γνώριζα από την αρχή ότι θα είναι δύσκολη η ψηφοφορία και ήμουν διατεθειμένη να προχωρήσω έστω και εάν δεν περνούσαν οι περισσότερες τροπολογίες που στοχεύουν στο να γίνει πιο φιλόδοξο το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα καταφέραμε όμως τώρα και μειώσαμε τις φιλοδοξίες του σχεδίου της Επιτροπής. Νομίζω όμως ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η πρόταση της ε, Επιτροπής που θα ήθελα να προτείνω στην ομάδα μου εν τέλει να απόσχει, ίσως και άλλες ομάδες να το προτιμήσουν αυτό. γιατί όσοι προτιμούν να φορολογούνται περισσότερο προϊόντα ενέργειας τα οποία είναι ρηπογόνα από την εργασία, αυτοί θα πρέπει να ξανασκεφτούν να είναι η πρόταση αυτή είναι σωστή. Ευχαριστώ κυρία Βαν Μπρέμπτ. Ψηφίζουμε τώρα το τελικό κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίας. 28 υπέρ. 16 κατά και 19 αποχές. Η επόμενη έκθεση που θα ψηφιστεί Η πρωτοβουλία για την πράσινη ζώνη. Εδώ έχουμε μόνο μία ψηφοφορία ε, με αποτέλεσμα υπέρ, κατά η αποχή και θα ζητήσω να σηκώσετε το χέρι. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται αυτή. Davis, Chris Davis, έχει το λόγο ως εισηγητής. Ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Θέλω να ελέγξετε τους αριθμούς των μελών των ομάδων. Ο πρόεδρος σε κάθε ψηφοφορία που διεξάγεται ηλεκτρονικά αυτομάτως ελέγχεται ο αριθμός και εγώ ανακοινώνω το εάν είναι παραπάνω από τα επιτρεπόμενα μέλη. Εάν υπάρχει αβεβαιότητα τότε να ζητήσετε ονομαστική, δηλαδή ηλεκτρονική ψηφοφορία, οπότε αυτομάτως εξασφαλίζεται ο σωστός αριθμός ψήφων κάθε πολιτικής ομάδας έχω μια ανακοίνωση ακόμη ότι η ενοποιημένη τροπολογία 17 αντικαθιστά, μάλλον περιλαμβάνει την τροπολογία 119. 109 διορθώνει ο πρόεδρος, 109 του κυρίου Σκυλακάκη. Αυτή έχει ενταχθεί στην υπαριθμόν 17 ενοποιημένη τροπολογία. Θα αρχίσουμε λοιπόν με την υπαριθμόν 1, ψήφι υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 2 συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παριθμόν 5 συμβαστική τροπολογία πάντοτε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή ακολουθεί η παριθμόν 17 όπου περιλαμβάνεται τώρα και η 109 υπέρ Κατά. Αποχές. Αυτή προτιμώ να την επαληθεύσουμε. Ψήφι υπέρ, όπως γνωρίζετε το σύστημα. ένα μέλος παραπάνω, σημειώνω, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Πέρας 34 υπέρ, 29 κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 6 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμών 7 συμβαστική υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και αυτή συμβαστική 8 υπέρ, κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμών 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική, ή μάλλον ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 10. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 11. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία μόνο 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 14 υπέρ κατά αποχές. Παρακαλώ να γίνει επαλήθευση. Ενωποιημένη τροπολογία 14. Πέρας. Υπέρ 30 και κατά 33, άρα απορρίπτεται. Ενωποιημένη τροπολογία 15, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε σε επιμέρους τροπολογίες τώρα. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα, ήτρε 1β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται αυτή. Τώρα, η 45, εδώ προβλέπεται κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Ας γίνει επαλήθευση. 45, τμήμα πρώτο. Πέρα τη ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 31 κατά. Άρα απορρίπτεται. Τότε. Ναι, με συγχωρείτε. Διότι, συγγνώμη, εκπίπτει ολόκληρη η τροπολογία. 46 και εδώ ζητείτε κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Α, το δεύτερο εκπίπτει λοιπόν και αυτό. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας γίνει παρακαλώ επαλήθευση. Die 38 υπέρ 24 κατά, ουδε μία αποχή, εγκρίνεται. Η παραδειθμόν 47 πρώτο μέρος, υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος εκπίπτει, ήτρε 5 υπέρ, κατά, αποχές, Παρακαλώ να γίνει επαλήθευση. Πέρας. 61 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Παρακαλώ να σηκώνετε καλά τα χέρια ώστε να μην είναι απαραίτητο να γίνεται η ηλεκτρονική επαλήθευση. 49 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 50 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 αποχές προτιμώ να προχωρήσουμε σε επαλήθευση υπέρ Α, νομίζω μάλλον ψηφίζουμε ηλεκτρονικά πέρας 52 υπέρ 10 κατά θα μας διευκολύνει να σηκώνετε καλά τα χέρια το δεύτερο μέρος υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτό. Ωραία, επαλήθευση του δεύτερου μέρους. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. 32 υπέρ, 30 κατά. Εγκρίνεται επομένως. 34 υπέρ. Α, με συγχωρείτε. Ναι, ναι, πρώτα την Άγκρη 2. Και αυτή σε δύο τμήματα, υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά, αποχές, εγκρίνεται δεύτερο μέρος, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Επαλήθευση για το δεύτερο μέρος της Άγκρη 2. Πέρας. 34 υπέρ και 29 κατά εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές. Αυτή απορρίπτεται. Ήτρε 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και ήτρε 21 δεν απαιτείται εδώ ψηφοφορία. Τώρα είμαστε στην ήτρε 4β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4γ 4σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές δεν είναι απόλυτα σαφές το αποτέλεσμα ας επαληθεύσουμε Πέρας. 32 υπέρ. 28 κατά. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Προτιμώ να κάνουμε επαλήθευση. 73. πέραστη ψήφου 30. Μία ψήφη υπέρ 29 κατά. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Καλώς. Επαλήθευση λοιπόν, 76. Πέρας. 30 υπέρ, 30 κατά. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Επαλήθευση δηλαδή. 93 λοιπόν. Πέρας. 31 υπέρ, 30 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση λοιπόν. 99. Πέρας. 30 υπέρ και 32 κατά απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κύριε Ντέιβις. Την 109. Α, έχει καλυφθεί, ναι. gehen jetzt weiter in der Abstimmung zu 100. 117 ακολουθεί τώρα. Ja, wir können 116 noch. Αν θέλετε να επαληθεύσουμε την ψηφοφορία της 116. Πέρας. 45 υπέρ, 8 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. 117, 118 και 119 και 20 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτονται. 121 υπέρ, κατά. Αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Ας κάνουμε παρήθευση. 122. Πέρας. 38 υπέρ και 24 κατά. Εγκρίνεται. 123 αυτή έχει αποσυρθεί. Η 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126. Α, αυτή εκπίπτει 126. 129 υπέρ κατά σχεδόν κανείς δεν σήκωσε το χέρι ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν 129 Πέρασε. 54 υπέρ 9 κατά. Παρακαλώ, σηκώστε καλά τα χέρια, γιατί θα μας διευκολύνετε πολύ. 131, Davis υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά μικρή πλειοψηφία υπέρ 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 Davis και Λίζε σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά εγκρίνεται θέλετε επαλήθευση δεύτερο τμήμα λοιπόν της 134-135 η, η ψηφοφορία έχει αρχίσει πέρας 37 υπέρ 26 κατά εγκρίνεται λοιπόν και αυτό 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή. Α, θέλετε λοιπόν επαλήθευση. Καλώς. Πέρας. 32 υπέρ. 30. Κατά. Συγχαρητήρια, αγαπητέ Κρίση. 137. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται και αυτή 140 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται το 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά, αποχές, ας το ελέγξουμε. 142 τροπολογία. Πέραση της ψηφοφορίας. 38 ψήφοι υπέρ, 25 κατά. Επομένως εγκρίνεται η τροπολογία αυτή. Τροπολογία 143 και 144 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτονται. 145 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτονται. 146 υπέρ, κατά. Ελέγχουμε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 απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτρε 20α δεν χρειάζεται να τις ψηφίσουμε ψηφίζουμε το 20β όμως της Ήτρε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προϊόν 155 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 156. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε θέλετε. Πέρας ψηφοφορίας. 33 υπέρ 28 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. 158. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 159 και 60. 100 και 160 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 162. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές και αυτό εγκρίνεται. Ας το ελέγξουμε. Εντάξει, δεύτερο τμήμα, έλεγχος της 162. Πέραση ψηφοφορίας. 34 ψήφοι υπέρ, 30 κατά. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα λοιπόν. Πηγαίνουμε στα 163 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι Κατά. Υπέρ λέω το πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ήτρε 15. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. δεν είναι σαφές. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ της 165. Κατά. Απορρίπτεται. Ήτρ... Να, ας το ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 165. Πέρας ψηφοφορίας. 38 ψήφοι υπέρ, 25 κατά. Εγκρίνεται. Η 8, δεν ψηφίζουμε. Τρόπο 166 ούτε και εδώ ψηφίζουμε. Ούτε και στη 10α. Αλλά η 10β ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρα, περνάμε στην άγκρη 5, στην άλλη σελίδα υπέρ, κατά, Επαναλαμβάνω. Ψήφι υπέρ, άγκρι 5. Κατά. Εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ήτρε 13 δεν ψηφίζουμε. Τροπολογία 180. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε, εντάξει. Πρώτο τμήμα της 180. Πέραση ψηφοφορίας. Ισοψηφία 29 υπέρ 29 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίσουμε κατευθείαν, λέω, με τα μηχανήματα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 47 ψήφοι υπέρ, 15 κατά. 181 του Ντέβις υπέρ, κατά, δεν είναι ξεκάθαρο. Ποιοι είναι υπέρ, σε 182 λέει τώρα ο Πρόεδρος. Ήτρε 14 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Άγκρι 16 υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. 17 άγκρι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 20 δεν ψηφίζουμε. Άγκρι 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 16 δεν ψηφίζουμε. 183 υπέρ, κατά. Φαίνεται να έχει απορριφθεί. Πηγαίνουμε στην άκρη 24. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 11, δεν ψηφίζουμε. ...189 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο, καταπίπτει. 190 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να ελέγξουμε. Την 190. Πέρας ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 30 κατά, Επομένως, απορρίπτεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 206 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 208 Ελέγχουμε την 207. Καλώς. Ελέγχουμε την 207. Πέρας ψηφοφορίας. 32 ψήφοι υπέρ, 31 κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογική 208. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε και την 208. Πέρας. 31 όλα. Απορρίπτεται επόμενος. 209 υπέρ. Δεν λειτουργήσε το μηχάνημά μου. Α, δυστυχώς αργήσατε να μας το πείτε. Λοιπόν, 209 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Άγκρη 19 υπέρ. Chris. Μας είπατε ότι άργησε να ψηφίσει. Μα δεν ήταν αυτό το θέμα. Ε, το μηχάνημα δεν λειτουργήσε. Δεν ήταν ότι άργησε. Ε, τι απόφαση πήρε τελικά εδώ. Κρίς, απλά είχα ε, κηρύξει το πέρας της συγκεκριμένης ψηφοφορίας. Αυτό εννοούσα. Τι θα πει πέρας ψηφοφορίας. Και είχα μάλιστα εκφωνήσει και το αποτέλεσμα. Ναι, αλλά η συνάδελφος μετά είπε ότι ψήφισα και δεν ε, λήφθη υπόψη ψήφος μου. Πρόεδρος, δηλαδή πόση ώρα πρέπει να διαρκεί κάθε ψηφοφορία. Έχουμε ψηφίσει και ο σχηρός και με, το μηχάνημα. Τώρα, αν κάποιος δεν έχει ψηφίσει ή άργησε ή δεν του αρέσει το αποτέλεσμα, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Ήταν σαφές κατά την άποψή μου. Όχι, δεν ήταν σαφές, λέει ο κύριος Ντέβις γιατί ήταν ε, τσίμα-τσίμα. Εγώ θα πρώτα να ψηφίσουμε. Λοιπόν, ο πρόεδρος όχι, ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Μπορεί να μην ήταν πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Όχι, δεν ήταν μικρή διαφορά. Ήταν 32 όλα νομίζω. Υπέρ... Θέλετε να το επαναλάβουμε. Μα αφού έχει απορριφθεί. Δεν θέλω να ξαναψηφίσουμε ηλεκτρονικά, λέει ο πρόεδρος. Είναι σαφές. Είχα κλείσει την ψηφοφορία. Και μετά έδωσε και το αποτέλεσμα. Δυστυχώς, λυπούμε, αλλά την επόμενη φορά που θα χρειαστεί, παρακαλώ να ζητήσετε τον λόγο έγκαιρα. Επέτρεψα αρκετό χρόνο για την ε, ε, ψηφοφορία. Τώρα, η Άγκρη 19, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 210. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 2.13 έχει αποσυρθεί. 2.14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.16 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, 217 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 218 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 219 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται 221 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 222 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 223 και κάποιες ακόμα είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. να ελέγξουμε τους 23, 24, 25. Der Wahlgang wird in Sekunden geschlossen. Und hier... Λοιπόν, πέρας της ψηφοφορίας. 33 ψήφοι πέρ, 30 κατά εγκρίνονται. 233. Περνάμε λοιπόν τώρα στην τροπολογία πρώτη, 2.33 υπέρ, κατά, αποχές, από 2.34 υπέρ, κατά, αποχές, ήτρε 9. Συγγνώμη, 235 λέει ο πρόεδρο. Υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 9 δεν ψηφίζουμε. 236. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 237. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 238. Υπέρ. Κατά. αποχές ελέγχουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 34 ψήφοι πέρα 27 κατά. 239, γιατί 17 ήταν δεν την ψηφίζουν. 239 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 241 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 240 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 240. Der Wahlgang ist jetzt geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. 34 ψήφοι υπέρ, 26 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογή 242 υπέρ, κατά. Αποχές. Παρακαλώ να ψηφίζετε ή να σκόντε τα χέρια σας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 243 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ελέγχουμε, ελέγχουμε, το 243. Πέρας. 48 υπέρ 12 κατά δεν υπάρχουν αποχές, εγκρίνεται. 244 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 246 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 247 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 245 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 248 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 250 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 249 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Όχι, ελέγχουμε, εντάξει. Με τα 249. Abstimmung ist Πέρας ψηφοφορίας. 33 ψήφοι υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 251 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Να σκόνετε καλά τα χέρια. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Εγκρίνεται τώρα. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 257 και 258. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 259, 260. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 261 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 262 και 263. Α, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 264-265. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ήτρε 12 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 266 δύο τμήματα πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται και αυτό. 267. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 268. Τρία τμήματα έχουμε εδώ. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά άποχες και αυτό εγκρίνεται. 269 ψήφι υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 270 υπέρ. Θέλετε τι, να ελέγξουμε το 269, καλώς, ελέγχουμε λοιπόν. Κατά, λέει ο πρόεδρος. Δεν έχω μπερδευτεί. Πέρας ψηφοφορίας, 23 ψήφοι υπέρ, 36 κατά απορρίπτεται. 2,70 υπέρ, κατά, αποχές. Ούτε και αυτό μου φαίνεται ξεκάθαρο. Ας ελέγξουμε και το 270. Πέρας ψηφοφορίας. 49 υπέρ 12 κατά εγκρίνεται 270. Επόμενη τροπολογία 281 υπέρ. ...281. Η 14 δεν εγκρίθηκε, άρα πρέπει να ψηφίσουμε την 281. Υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. Εντάξει, ελέγχουμε, ελέγχουμε την 281. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 33 ψήφοι υπέρ, 27 κατά. Επόμενη, άγκρι 1. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Άγκρι 9 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 10 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Καλά, ας την ελέγξουμε. Άγκρι 10. Πέρας ψηφοφορίας. 38 υπέρ 23 κατά. Εγκρίνεται. Άγκρι 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 282 υπέρ. 282 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 11 υπέρ. Κατά. Αποχές Ναι, σαφέ. σαφές. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 11 τη Επιτροπής Γεωργίας. Πέραση ψηφοφορία. Σαφέ ήταν, αλλά εγώ δεν έβλεπα από εδώ, λέει ο πρόεδρο. 54 ψήφοι υπέρ, 6 κατά. Άγκρι 12 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Άγκρι 14 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Εγώ θα ήθελα να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. Πέραση ψηφοφορίας Εγκρίνεται 36 υπέρ 23 κατά. Άγκρι 21 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη σι 1C1 γάμα. Ε, δεν την ψηφίζουμε, όχι. Industry 2. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τρεπτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 294 ψήφι υπέρ κατά αποχές νομίζω ας, ας επαληθεύσουμε άλλη μια φορά φαίνεται πάντως να εγκρίνεται επαλήθευση 294 Abstimmung ist geschlossen. Πέρας της ψηφοφορίας 32 υπέρ 29 κατά δεκτή. Δύο 95-96 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτές. 97 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 298 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22α ήτρε δεν θα ψηφιστεί. 299 πλέον και είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ήτρε 22β μικρό. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 22β μικρό ήτρε. Πέρας της 39 υπέρ, 14 κατά δεκτή. 19 ήτρε ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην 307 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η 307. 308 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 309 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 310 υπέρ, κατά, αποχές, δεν έχει διευκρινιστεί. γιατί την 310 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας 29 υπέρ 31 κατά απορρίπτεται. 311 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 312 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 313 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεν θα πρέπει να ψηφίσουμε την 314 Περνάω στην 315 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 316 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 317 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τοπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τοπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τοπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τοπολογία 5 και 6 ταυτόσημες υπέρ. Κατά Αποχές δεν έχει διευκρινιστεί. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 5 και 6 μαζί. Πέρα στις ψηφοφορίες. 27 υπέρ, 33 κατά απορρίπτεται. Περνάμε στην 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές. Επαναλαμβάνουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος ζητείτε λοιπόν για την 8. Ξεκινάμε. Τέλος της ψηφοφορίας. 33 υπέρ 27 κατά. Δεκτή. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 12 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 13 υπέρ. Συγγνώμη, καταπίτη. Η 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 15, παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 35 κατά, απορρίπτεται. 16 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, δε, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή ηλεκτρονικός έλεγχος και για τη 17 να είμαστε σίγουροι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 27 υπέρ, 33 κατά απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Σε δύο τμήματα μάλλον. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 22. Ψηφίζεται. Πέραση ψηφοφορίας. 32 υπέρ 28 κατά δεκτό το δεύτερο τμήμα. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ καταπίπτει 25. 26 υπέρ κατά απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές από ό,τι φαίνεται δεκτή 32 υπέρ κατά αποχές η ξανά υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή 32, η 30 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ο Κρίς. Ξέρουμε ότι υπάρχει και άλλη μια σημαντική ψηφοφορία. Το θέμα είναι αν θα προλάβουμε να το κάνουμε γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Thank um, Due to the several new um, limitations, conditions and targets, I would like to suggest... Σχετικά με τους νέου περιορισμούς που τέθηκαν, θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να καταψηφίσουν την έκθεση, λέει η κυρία Σίζελη. Ζητάτε μια διακοπή, κύριε Ντέιβις. υπάρχει κάποιος χρόνος για μια πάρα πολύ μικρή ε, ε, διακοπή. Πέντε λεπτά διακοπή. Θα προλάβουμε να κάνουμε και την επόμενη έκθεση. Κοιτάξτε, βλέποντας την ώρα η οποία έχει προχωρήσει, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε την έκθεση χάση, αυτό είναι δύσκολο. Λοιπόν, πέντε λεπτά διακοπή. Πρόεδρε, νομίζω ότι έχει σημασία να ψηφίσουμε και τη δική μου έκθεση σήμερα. Αν οι ομάδες έχουν ανάγκη για χρόνο, μπορούν να το κάνουν αυτό κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας της εκθεσιός μου. Λοιπόν, να ψηφίσουμε τη δική μου έκθεση και να ψηφίσουμε την τελική ψήφο για την προηγούμενη έκθεση μετά το τέλος της δικής μου. Δεν ξέρω γιατί έγιναν οι αλλαγές αυτές ε, ε, στην ε, ημερήσια διάταξη, προφανώς λόγω των προβλημάτων με τις πτήσεις χθες. Καταφέραμε όμως να είμαστε όλοι εδώ σήμερα και ακόμα και αν ξεπεράσουμε το χρόνο μας δεν πειράζει, ας ψηφίσουμε. Αυτό που δεν γίνεται με κανένα τρόπο είναι να αναμίξουμε τις δύο ψηφοφορίες. Βρισκόμαστε τώρα στην ψηφοφορία του κυρίου Ντέιβις, της εκθέσεως Ντέιβις. Και ω εισηγητή, ο κύριο Ντέιβι ζήτησε διακοπή πέντε λεπτών για να μπορέσει να διαβουλευτεί. Γιατί η έκθεση είναι σημαντική και διότι πρόκειται να μπούμε στην τελική ψηφοφορία και ε, επιθυμούν να συζητήσουν τι στάση θα κρατήσουν. Παρακαλώ λοιπόν να εγκρίνουμε τα πέντε λεπτά διακοπή που ζητεί ο κύριος Ντέιβις και μετά θα προχωρήσουμε στην επόμενη ε, ψηφοφορία. Θα συζητήσουμε την περαιτέρω διαδικασία και στο διάλειμμα μπορούν να συζητήσουν οι συντονιστές τι ακριβώς θέλουν να πράξουν. Διακοπή λοιπόν για πέντε λεπτά. Στις 12 και 25 συνεχίζουμε. Ο πρόεδρος, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πέρασαν αυτά τα πέντε λεπτά. Σας παρακαλώ καθίστε. Καλά λοιπόν, βρισκόμαστε ακόμη στην ψηφοφορία της εκθέσεως Davis και προβλέπεται τώρα η τελική ψηφοφορία. Αυτή θα γίνει ονομαστικά, δηλαδή ηλεκτρονικά. Ψηφίστε λοιπόν αν θέλετε. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Εδώ πέρα τούτε η ψηφοφορία. 32 υπέρ, 24 ψηφι κατά και 5 αποχές. Άρα συγχαρητήρια στον κύριο Ντέιβις και προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή τα ναυτικά καύσιμα. Και εδώ παρακαλώ σύντομα να δηλώσουν οι συντονιστές με ποιον τρόπο επιθυμούν να χειριστούμε την ψηφοφορία αυτή. Έχουμε το πολύ 10 λεπτά με διερμηνία. Όμως η ψηφοφορία προβλέπω ότι θα κρατήσει τουλάχιστον 30 λεπτά, άρα χωρίς ψηφοφορία πλέον, χωρίς ε, διερμηνία σύγχρονη πλέον. Θα προτείνω λοιπόν δεν ξέρω ποιο είναι ο αρμόδιο συντονιστή του Λαϊκού Κόμματο, ο κύριο Ζέμπερ. Ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε. Είναι θλιβερό το αποτέλεσμα κατά την άποψή μου, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή. Εφόσον δεν θα είναι διαθέσιμη η διερμηνία μετά από 10 λεπτά, θα είναι δύσκολο να γίνει ψηφοφορία. Προτείνω και η ομάδα μου ζητεί την αναβολή. Λίντα Μακάβανε. Η ομάδα μου ψηφίζει ευχαρίστως και τώρα και χωρίς διερμηνία. Κύριε Ντέιβις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κύριος Ζέμπερ έχει δίκιο. Ψηφίζουμε νομοθετικό κείμενο και οφείλουμε να τηρούμε τους κανονισμούς και οι κανονισμοί προβλέπουν διερμηνία. Σα του χάσει. Εγώ επισημαίνω, αν εξετάσετε την, λίστα ψηφοφορίας, θα δείτε ότι όλα σχεδόν καλύπτονται με ε, τροπολογίες συμβιβαστικέ ή ενοποιημένε, που σημαίνει ότι η ενοποιημενε που σημαινει οτι η φοφορια δεν θα κρατήσει μισή ώρα. Ελπίζω να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τώρα, διότι πρόκειται για νομοθετικό ζήτημα και οι ενδιαφερόμενοι ζητούν, χρειάζονται την βεβαιότητα, χρειάζονται την ασφάλεια. Το ECR. Δεν μας ικανοποιεί η προοπτική αναβολής, αλλά οι κανονισμοί είναι κανονισμοί και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή λύση. Εσείς υποστηρίζω την εισηγήτρια να ψηφίσουμε τώρα δηλαδή. Ο κύριος Ρώση. Είμαστε υπέρ του σεβασμού των κανόνων. Βλέπω ότι έγινε και άλλη μια ανακοίνωση στους συντανάστρους. Δεν ξέρω τι γίνεται ε, σε σχέση με την αποζημίωση των διερμηνέων. Έτσι κι αλλιώς ε, δεν βλέπω. Εφόσον πληρώνονται για όλη την ημέρα, ποια είναι το πρόβλημα να δουλέψουν άλλη μισή ώρα παραπάνω, λέει ο κύριος Ρώση. Εσείς κύριε συνάδελφε, επί του διαδικαστικού. Για διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση που είναι πολύ σημαντική νομοθετική πρόταση και που θα επηρεάσει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και τις δουλειές τους δεν έχει, δηλαδή οι τροπολογίες επί της εκθέσεως, οι αρχικές τροπολογίες δεν έχουν συζητηθεί. Εγώ ήλεγξα τις ημερήσεις διατάξεις, οι Τροπολογίε κατατέθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου και δεν υπήρξε η δυνατότητα, δεν υπήρξε η ευκαιρία να συζητηθούν. Είναι λοιπόν το νόμιμο δικαίωμα καθενός συναδέλφου να υποστηρίξει τις τροπολογίες του. Εάν δεν διεξαχθεί συζήτηση για τις τροπολογίες σε νομοθετική έκθεση, μα τότε τι θα συζητήσουμε. Νομίζω ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε στους συναδέλφους την δυνατότητα, εγώ ο ίδιος θέλω να υποστηρίξω τις τροπολογίες μου και έχω το δικαίωμα αυτό, να συζητήσουμε λοιπόν τις τροπολογίες σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις και μετά να προχωρήσουμε σε μία ορθή ψηφοφορία. Ας μην ψηφίζουμε χωρίς συζήτηση. Ο πρόεδρος, άκουσα όλες τις απόψεις. Κύριε Ρώση, Ε, ο κανονισμός προβλέπει διερμηνία για τις συζητήσεις, όχι απαραίτητα για τις ψηφοφορίες, δεν το λέει αυτός ο κανονισμός. Αλλά για να είναι σοβαρή η επεξεργασία του φακέλου, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να, προβλέπει, να υπάρχει και διερμηνία. Προτιμώ λοιπόν να αναβάλουμε για μια από τις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ένβη. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δυσάρεστο αυτό, αλλά για να είμαστε πραγματικά σοβαροί, παρακαλώ να δεχτείτε αναβολή. Οτιδήποτε άλλο δεν θα ήταν σοβαρό, διότι υπάρχουν πολλέ επιφυλάξεις από πολλούς. Η γραμματεία μου λέει ότι θα χρειαστούμε το λιγότερο 30 λεπτά. Θα διαμορφωθούν λοιπόν συμπτωματικές πλειοψηφίες και για την κυρία Χάση θα πω ότι αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες, ορισμένες από αυτές, δεν, δεν βασίζονται σε πολύ στέρεο έδαφος. Γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλέσω όλες και όλους να συμφωνήσετε να ε, αναβληθεί η ψηφοφορία. του Χάση. Εάν αυτή είναι η γνώμη της πλειοψηφίας δεν μπορώ να αντιταχθώ. Ελπίζω όμως στο Στρασβούργο να μπορέσει να διεξαχθεί έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής για να διεξαχθεί αυτή η ψηφοφορία καθώς επίσης για να γίνουν και σχόλια επί των τροπολογιών. Η ίδια ψηφοφορία δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο διότι σχεδόν όλα καλύπτονται τώρα με όπως είπα συμβαστικές ή ενοποιημένες τροπολογίες. Ο Πρόεδρος Πέμπτη πρωί στο Στρασβούργο νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να διεξαχθεί η ψηφοφορία και μπορώ να σας υποσχεθώ ότι στο μέλλον σήμερα συζητήσαμε δύο θέματα που μας πήραν πολύ χρόνο. Στο μέλλον, παρακαλώ, παρακαλώ, χαρίστε μου την προσοχή σας ακόμα για λίγο. Στην συνάντηση των συντονιστών θα συζητήσουμε έτσι ώστε η ψηφοφορίες επί νομοθετικών προτάσεων να έχουν προτεραιότητα και να γίνεται και η απαραίτητη συζήτηση. Και απευθύνομαι τώρα και στους σκιώδεις συγητές. Να λάβετε υπόψη σας ότι και οι σκιώδεις συγητές, σαν του Χάση, σε σας απευθύνομαι, να έχουν τη δυνατότητα να συζητούν και τις τροπολογίες. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο για να υπάρχει σεβασμός των απόψεων. Και όπως είπα, πέμπτη πρωί νομίζω θα μπορέσει να γίνει η ψηφοφορία καθώς επίσης και η συζήτηση που ζητήθηκε από πολλές και πολλούς συναδέλφους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εύχομαι καλό μεσημεριανό διάλειμμα και θα σας δω στο Στρασβούργο. Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ασφαλιστεί η διεξαγωγή της ψηφοφορίας εκεί.